So. So, ladies and gentlemen. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, οι διερμηνείς σας ενημερώνουν ότι βρισκόμαστε στην 30η μέρα των κινητοποιήσεών μας και και διαμάχη με τη δίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά συνέπεια δεν θα παραχωρήσουμε σήμερα υπέρβαση ωραρίου και η διερμηνία, θα σταματήσει στις 4.30 ακριβώς. Ladies και κύριοι, Uh, Καλώς ορίσατε σε αυτή την κοινή συνεδρίαση. Ντεβε και Άφετ. Η ε, κυρία Μακάγουαν και εγώ σας υποδεχόμεθα με χαρά όλους. Είμαστε στο σημείο 1. Έγκριση ημερησίας διατάξεως. Μόνο ένα σημείο στην κοινή συνεδρίαση ΑΦΕΤ, του διευρυμένου Προεδρίου ε, της ΑΦΕΤ και των συντονιστών της ΔΕΒΕ η παρουσίαση του εξωτερικού χρηματοδοτικού μέσου περίοδος 2021-2027 Συμφωνείτε? Ωραία. Οπότε πάμε στο σημείο 2, ανακοινώσει του Προέδρου. Πέρα από τους ε, συντονιστές και αντιπροέδρους των Επιτροπών και της ε, Υποεπιτροπής ε, ΔΟΑ που συμμετέχουν και οι συγκεκριτές που εξετάζουν το θέμα της εφαρμογής των εξωτερικών χρηματοστατικών σημείων, Ενρίκο Γκερέρα και Σάκε, Ξεκινά η συνεδρίαση που είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη. Έχουμε γερμανικά, αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά, ολλανδικά, ελληνικά, ισπανικά, πολωνικά σε διερμηνία. Πριν δώσω το λόγο στη Λίντα Μακάβουν να κολοσορίσω την είπατε εκπρόσωπο και την πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη και τον επίτροπο Μιμιτσά. Αυτά και μπορεί να συνεχίσει Λίντα. Θα είμαι πολύ σύντομη, διότι οι διερμηνεί θα σταματήσουν ακριβώ στι 4.30 να καλωσορίσω όλους τους συναδέλφους. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε προτάσεις για τον, ε, τα νέα μέσα εξωτερικής δράσης πριν από 15 μέρες, 12 ε, χρηματοδοτικά μέσα που συναθρίζουν τα μέσα που εμπίπτουν σε αρμοδιότητες αντιστοίχων επιτροπών μας στα πλαίσια τη Επιτροπή Ανάπτυξη και Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, να ενημερώσω του επιτρόπου μα, λέγοντα ότι το Κοινοβούλιο μα πιθανότατα θα ακυρώσει αύριο απόφαση των ε, Προέδρων των Επιτροπών και θα υπάρξει μια επίσημη κοινή διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τις δύο Επιτροπές για αυτά τα μέσα και θα διορίσει η Επιτροπή μας ε, εισηγητές ε, την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, οι Επιτροπές μας μάλλον εισηγητέ. και μετά θα δεξαχθεί κάποιο συντονισμό συγγνώμη, για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βρούμε κοινή μέθοδο εργασίας και να καθορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το έργο μας. Χρειάζεται δύο να χορέψουν, ε, όχι μόνο με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θα θέλαμε να ξέρουμε πώς κινείται το Συμβούλιο. Έχουν θέσει κάποια ζητήματα, σας έχουν θέσει κάποια ζητήματα συνάδελφοι από πλευρά αναπτυξιακής. Μία από τις σημαντικότερες ανησυχίες μας είναι αυτό που λείπει από τους βασικούς στόχους. Είναι η εξάλληψη της φτώχειας, ε, που είναι βασική λειτουργία σύμφωνα τη συνθήκη των αναπτυξιακών αυτών μέσων και έχουμε και τους στόχους της χιλιετίας που έχουν τεθεί. Εντάσσεται αυτό και ξέρω ότι το υποστηρίζετε αυτό. Το είδα ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίση συμφώνησε ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη συνεχούς αναπτυξιακής βοηθείας και μάλιστα αυξήσεως αυτής και θα ήθελα να δω πώς αυτό θα αντικατοπτριστεί στα μέσα μας όπως θα, προχωρούμε. Το Κοινοβούλιο και οι συνάδελφοι θα το θέσουν το θέμα. Θεωρούμε ότι η πρόταση για περισσότερο έλεγχο ε, πρέπει να προβληθεί και χρειάζεται όμως και ταυτόχρονα μεγαλύτερη ευελιξία που σημαίνει ότι χρειάζεται όμως ο κατάλληλος κοινοβουλευτικός ε, έλεγχος, διότι εμεί λογοδοτούμε στους πολίτες μας για τη χρήση των πόρων και αυτό θα το συζητήσουν ε, εκτενώς οι ασχολούμενοι με το θέμα. Ε, αμέσως λοιπόν να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Δεν ξέρω αν David έχει να πει κάτι άλλο. Λοιπόν, ας δώσουμε το λόγο στην είπατε εκπρόσωπο να προχωρήσουμε, να είμαστε αποτελεσματικοί λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη Φεντερίκα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Λίντα, ευχαριστώ όλους για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας ε, παρουσιάσω την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα μιλήσω εκ μέρους του ε, Συμβουλίου για το νέο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα γνωρίζετε ότι ο Επίτροπος Χάν ήθελε να είναι εδώ σήμερα, αλλά ε, σας έγραψε μια επιστολή ε, να ε, εξέφρασε τη διαθεσιμότητά του να σας συναντήσει κάποια άλλη στιγμή γιατί δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Θα θυμάστε ότι είχαμε την πρώτη ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων και πριν από την έγκριση της πρότασης ε, σε άλλη αίθουσα, στο ίδιο κτίριο, τώρα που ε, οι νομοθετικές προτάσεις για τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα έχουν εγκριθεί. Μπορούμε να αρχίσουμε να συζητούμε τις λεπτομέρειες. Ξέρω ότι ο Νέβεν θα, σας αναφέρει άλλα στοιχεία ε, που απασχολούν όλος ιδιαίτερο στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Ε, θα ήθελα λοιπόν εγώ να σας παρουσιάσω τη γενική προσέγγιση, τα πιο γενικά ε, στοιχεία. Κάτι που δεν πρέπει να μας διαφεύγει είναι ότι η πρότασή μας ε, συμπεριλαμβάνει μία αύξηση της τάξης 30% του προπολογισμού για τα εξωτερικά μέσα. Διπλό είναι το μήνυμά μας. Πρώτον, γιατί η δουλειά μας ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός συνόρων είναι πάρα πολύ σημαντική και για τους πολίτες και για ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπουμε όλο και περισσότερο δυνάμεις έχουν μια ε, τάση απόσυρσης ε, στην παγκόσμια σκηνή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποστέλει ένα μήνυμα με την αύξηση αυτή της εξωτερικής δράσης ε, ότι δεν αποσυρώμαστε από τις ευθύνες μας και από τα παγκόσμια δρόμενα αντιθέτω, θέλουμε να συμμετέχουμε ακόμη περισσότερα στην παγκόσμια, στο διεθνές προσκήνιο η δουλειά που έχουμε κάνει κατά τα τελευταία χρόνια έχει καρποφορήσει. Είναι η σωστή προσέγγιση για μια ε, εξωτερική πολιτική ε, κατάλληλη. Θέλουμε λίγο περισσότερες επενδύσεις όσον αφορά την εξωτερική πολιτική μας. Αυτό ζητούν οι εταίροι μας σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να σας πω ότι το μήνυμα αυτό έχει γίνει κατανοητό. Η υπηρεσία μας ε, συναντήθηκε με, τις, κυβερνητικές οργανώσεις και τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών ε, προσπαθήσαμε να του εξηγήσουμε ότι περισσότερα χρήματα δίνουμε για τις προτεραιότητες που είναι οι κοινέ μα προτεραιότητες, για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αηφόρο ανάπτυξη, την εξάλληψη της πτώχεια, ε, την ε, αντιμετώπιση κλιματική αλλαγή και για τη γειτονία αλλά και για την ανθρωπιστική βοήθεια. Θέλουμε να έχουμε καλύτερα εργαλεία για να μπορούμε να επενδύουμε στι προτεραιότητε μα, αλλά οι προτεραιότητε μα είναι σαφώ προκαθορισμένες και οι περισσότερε δεν αλλάζουν. Έχουμε αντιμετωπίσει καταστάσει κατά τι οποίε χρειάστηκε να προσαρμόσουμε τι πολιτικέ μα ε, στα εργαλεία μα και με την πρόταση αυτή προτείνουμε να ε, δράσουμε αντίστροφα, να θέσουμε τι προτεραιότητέ μα και να να προτείνουμε ε, οικονομικά μέσα που εξυπηρετούν αυτές τις ε, προτεραιότητες ε, που καθορίζονται σε πολιτικό επίπεδο. Να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι προτεραιότητες μας πρέπει να ενσωματωθούν στις προτάσεις μας και μπορώ να σας πω ότι και ο Νίβεν και εγώ έχουμε προσέξει όλος ιδιαιτέρως το στοιχείο αυτό. Όσον αφορά τώρα το μέσο συνεργασίας ε, για τη γειτονία, την ανάπτυξη είναι, ε, περιλαμβάνει 90 ε, δις σε ποσό, θα αντικαταστήσει 9 από τα προηγούμενα μέσα. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή η εξωτερική δράση έχει ένα δυσανάλογα υψηλό επίπεδο μικρών εργαλείων σε σχέση με άλλες πολιτικές, δηλαδή έχουμε μια πολύ, ένα πολύ κατακαιρματισμένο σύνολο μέσων σε σχέση με τους συναδέλφους μας. Έχουμε λοιπόν επί καθημερινής βάσεως να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, δυσκολίες ε, που αντιμετωπίζουν οι εταίροι μας προσπαθώντας να, να αναγνωρίσουν ποιο είναι το σωστό εργαλείο για ε, το κάθε πρόβλημα. Όχι μόνο οι χώρες εταίροι αλλά και οι εφαρμοστικοί οργανισμοί, οι οργανισμοί που εφαρμόζουν τις προτεραιότητες αυτές, όλοι ζητούν μεγαλύτερη απλοποίηση ε, γιατί το επίπεδο εφαρμογής είναι πραγματικά πάρα πολύ υψηλό. Ε, πιστεύω ότι έτσι θα βοηθηθούμε και εμεί, ε, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, ω προ τη διαχείριση και την υποπτία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο πιο κατακαιρματισμένα είναι τα οικονομικά μέσα, τόσο, πολύ, τόσο πιο μεγάλο είναι ο κίνδυνο να χαθεί ε, ένα κομμάτι του παζλ. Όσον αφορά του ε, ε, στόχου αηφόρου ανάπτυξη, ε, του έχουμε συμπεριλάβει και αυτού σε αυτό το νέο εργαλείο που προτείνουμε. Ε, μιλούμε λοιπόν για όλες τις πολιτικές που πηγαίνουν, σε μια πιο πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης, πολιτική προσέγγιση στις προτεραιότητες εξωτερικής δράσης, ε, μια αυτόματη αντίδραση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ζητήματα που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Ε, όλα αυτά λοιπόν αφορούν μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, όχι μεμονωμένη προσέγγιση που μερικές φορές έχουμε ακολουθήσει ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε στους θεσμούς μας. Η πρότασή μας για τον προπολογισμό λοιπόν πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Το νέο μέσο έχει διαμορφωθεί ε, στην ίδια λογική με την ατζέντα για το 2030 των Ηνωμένων Εθνών. Οι λεπτομέρειες τώρα ε, συνεργασίας μας ε, πρέπει να είναι διαφοροποιημένες για τις διαφοροποιημένες προτεραιότητες. Η πρόταση τη συμπεριλαμβάνει. Οι βέλτιστες πρακτικές θα συμπεριληφθούν στο νέο ε, μέσο. Επικεντρωνόμαστε σε κάποιες από τις προτεραιότητες. Πρώτον, η γειτονία. Πρόκειται για ένα μέσο για την γειτονία μας. Ε, η πρότασή μας ε, αυξάνεται κατά 25%, 22 δις ευρώ δηλαδή ε, και πιστεύω ότι δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρότερο μήνυμα της πολιτική μας γειτονίας και της ενίσχυσης συνεργασίας μας με τους προσανατολάς εταίρους μας αλλά και με τη Μεσόγειο και επίσης θα ορίσουμε τις ιδιαιτερότητες μαζί με τους εταίρους μας. Το νέο μέσο θα επικεντρώνεται στις επιδόσεις. 10% της χρηματοδότησης για την περιφέρεια θα εξαρτάται με την οικονομική διακυβέρνηση και την πρόοδο στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η υποστήριξη της περιφερειακής συνεργασίας είναι πάρα πολύ σημαντική επίσης ε, και στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης ε, και ε, της Μεσογείου και την περιφερειακή συνεργασία γύρω από τον Εύξηνο Πόντο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ξεπεράσουμε κάποια τεχνητά εμπόδια που έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία δύο χρόνια. Δύο παραδείγματα να σας δώσω που εμένα προσωπικά με σοκάρισαν από την καθημερινή μας εργασία. Η Μαυριτανία έχει τώρα προσχωρήσει στην Ένωση για τη Μεσόγειο, όμως δεν καλύπτεται από το τρέχον μέσο γειτονία και είχαμε και έχουμε προβλήματα χρηματοδότηση ε, έργων ε, με την Ένωση τη Μεσογείου ε, που αφορούν τη Μαυριτανία. Ε, γιατί πολλές φορές η πολιτική, ε, εξωτερική μας πολιτική πηγαίνει πέρα από τα μέσα που έχουμε εγκρίνει. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε αναπτύξει ένα πάρα πολύ ενεργό ε, δίκτυο, δραστήριο δίκτυο νέων ηγετών ε, Στι χώρε του Σεχέλ και στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκής, της Αφρικανικής Ένωσης και στη Μεσόγειο νέους ανθρώπους από το Ιράκ και το Περσικό κόλπο δεν μπορέσαμε να τους συμπεριλάβουμε γιατί δεν καλύπτονταν από το μέσο ε, αυτό. Είναι δίκαιο, είναι λογικό, είναι φυσιολογικό, μας βολεύει, όχι δεν μας βολεύει. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια τέτοια προσέγγιση που θα μας επιτρέπει, θα επιτρέπει στους ε, διαδόχους μας να χρησιμοποιήσουν τα μέσα αυτά με τις σαφείς πολιτικές προτεραιότητες αλλά με κάποια κάποια αλφα ευελιξία ε, που να ε, ε, εξηγείται από το γεγονός ότι ο κόσμος αλλάζει συνεχώς και είναι διαφορετικός από αυτόν που τον γνωρίζαμε. Έχουμε λοιπόν και ένα ξεχωριστό μέσο με αναγνώριση των υποψηφίων χωρών και της ειδική τους θέσης στην καθημερινή μας δουλειά, 13% αύξηση του συγκεκριμένου ταμείου για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερο τα Δυτικά Βαλκάνια όπως προχωρούν καθώς προχωρούν ε, στην ε, ε, προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το προενταξιακό μέσο λοιπόν θα συμπεριλάβει και τη σχέση μας με την Τουρκία ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουν, που υποστη... να υποστηρίξουμε αυτούς που υποστηρίζουν τις ευρωπαϊκές αξίες εντός της Τουρκίας. Το κάναμε και κατά τα τελευταία έτη. Αν θυμάμαι καλά, ο Επίτροπος Χάν ούτως ή άλλως σας είπε τα σχετικά τη ανταλλαγή αυτής απόψε, τελευταία φορά που, που συναντηθήκαμε που συναντηθήκατε. Εμείς προτείνουμε μια μεγαλύτερη δέσμευση για την αναπτυξιακή συνεργασία. Οι μακροχρόνιες προτεραιότητες δεν μπορούν λόγω της βραχυπρόθεσμης πίεσης να θυσιαστούν αηφόρο ανάπτυξη και σχετική στόχη, αηφόρο ε, ανάπτυξη με βασικό, ε, με βασικό στόχο η εξάλληψη τη φτώχεια. αυτό είναι σαφέ για μα. Όλοι γνωρίζουμε, ε, όσοι είμαστε εδώ στην αίθουσα, ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, έχουμε αντιμετωπίσει πιέσει να δώσουμε κάποια ποσά, να τα πάρουμε από αυτό το μέσο και να τα δώσουμε σε άλλε κρίσει. Αντισταθήκαμε σε αυτό πρέπει να πω, αλλά πιστεύαμε, πιστεύουμε ότι, να, ότι είναι λογικό να σκεφτούμε ότι η διάδοχή μα μα θα έχουν τέτοια προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό ακριβώ θέλουμε ένα αποθεματικό το οποίο θα αφιερωθεί σε αυτό ώστε να γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα ε, ποσά που θα φορούν τις μακροχρόνιες επενδύσεις πολιτικές μας και ούτω καθεξής ε, θα ε, θα έχουν ως αποτέλεσμα να αποφευχθεί αυτή η πίεση στο επόμενο κοινοβούλιο ή στην επόμενη επιτροπή ε, να ε, πάρουν τα ποσά αυτά και να τα δώσουν αλλού. Έχουμε λοιπόν ένα αποθεματικό για, για κατεπήγουσες καταστάσεις, κάτι που ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όταν χρειάστηκε να προωθήσουμε, να αυξήσουμε τις επενδύσεις μας στο Ταμείο για την Αφρική, την αντιμετώπιση του τυφώνα Ήρμα και άλλων θεομηνιών Αποφασίσαμε λοιπόν ε, να το κάνουμε αυτό για ολόκληρη την πρότασή μας. Τα αναπτυξιακά ποσά θα αφορούν μόνο μακροπρόθεσμα, ε, μακροπρόθεσμες ε, πολιτικές και προτεραιότητες. Όσον αφορά τώρα το μέσο διεθνού συνεργασίας για ζητήματα που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, 1,5 δις ευρώ για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας και και ακόμα 1,5 δις ευρώ για τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών οι λεπτομέρειε συνεργασία, τρόπο συνεργασία μα ε, που έχει λειτουργήσει καλά, έχει συμπεριληφθεί σε αυτή την πρόταση. Θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μα με τι ε, μη κυβερνητικέ ε, οργανώσει, οι οποίοι μα είπαν ότι μέχρι τώρα συμφωνούν με τις προτάσει μα. Αυτέ ήταν οι βασικέ προτεραιότητε που καλύπτουν τόσο ή άλλως από το προηγούμενο μέσο και που θα είναι τμήμα και του καινούριου μέσου. όμω η νέα πρόταση αντανακλά και κάποιε νέε προτεραιότητε προτεραιότητες και δεσμεύσεις ε, τις οποίες επεξεργαστήκαμε κατά τα τελευταία χρόνια. Πρώτα, το, πρώτα απ' όλα το κλίμα. Τουλάχιστον προτείναμε ε, να αντανακλάται αυτός ο φιλόδοξος στόχος σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό, 25% στόχος για την κλιματική αλλαγή. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα ε, όταν κάποιοι στον κόσμο φεύγουν από συμφωνίε όπω η Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, είναι σημαντικό να δώσουμε αυτό το μήνυμα ότι εμεί παραμένουμε δεσμευμένοι. Είναι και πολιτικό μήνυμα αυτό. Δεύτερον, μετανάστευση. Το νέο μέσο στοχεύει να συμπεριλάβει επίση επιμένω σε αυτό, να συμπεριλάβει, να ενσωματώσει τη μετανάστευση στι συμφωνίε με τους, στη συνεργασία με του εταίρου μα. Γιατί διαφορετικά θα κινηθούμε προ κατευθύνσει οι οποίε δεν συνάδουν υποχρεωτικά με τι αξίε μα, ε, τι αρχέ μα, ούτε με τη συνοχή των πολιτικών μα. Ε, θέλουμε συμπληρωματικότητα μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών μεταναστευτικών πολιτικών ε, και σύμφωνα με τα τελευταία συμπεράσματα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 10% αύξηση του, των δαπανών περίπου 9 δις ευρώ δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε και τις αιτίες της παράνομης μετανάστευσης και την υποχρεωτική τον υποχρεωτικό εκτοπισμό. Ε, αυτό θα καλύψει δηλαδή τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης, των πολιτικών μας για τη μετανάστευση και τέλος πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την αύξηση της ικανότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την πρόληψη συγκρούσεων στο εξωτερικό, διατήρηση της ε, ειρήνης, την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας. Θέλουμε μία ισχυρή ικανότητα για την πρόληψη των συγκρούσεων. Εγώ προτείνω μία, τη δημιουργία μια διευκολυνση για την ειρήνη εκτό προπολογισμού. Όλες τις δραστηριότητες στρατιωτικής φύσεως που είναι εκτός του προπολογισμού θα χρηματοδοτούμε έτσι ε, για να μπορέσει να υποστηρίξει τη δουλειά για την ασφάλεια και την άμυνα που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια. Πάλι θα χρειαστεί ένα ειδικό χρηματοδοτικό μέσο. Είναι εκτός προπολογισμού όμως ε, και δεν είναι τμήμα της ε, πρότασης ε, που έχετε μπροστά σα. Απλώς είναι στο ευρύτερο πλαίσιο της δουλειάς του, διεθνού, του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου ε, θα ήθελα να ολοκληρώσω με αυτό. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που καθυστέρησα και που μίλησα πολύ, αλλά πρέπει να πω ε, πριν ολοκληρώσω το εξή. Εσείς θα αποφασίσετε, ε, σας δίνουμε μεγαλύτερη δυνατότητα εποπτείας με τη νέα πρόταση, γιατί όπως σας είπα προτείνουμε παράταση των αρμοδιοτήτων, ε, επέκταση μάλλον των αρμοδιοτήτων ε, της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα που αφορούν ολόκληρο τον κόσμο και τις πολιτικές μας για τον ολόκληρο τον κόσμο. 30 δις επιπλέον δηλαδή θα είναι υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή όμως μια πρόταση πρόταση που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι που το έχετε ζητήσει πολύ καιρό. Ε, θα πρέπει βέβαια να γίνει δουλειά όταν θα περάσουμε στην διαδικασία λήψη αποφάσεων για τον προπολογισμό. Το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι είναι το σωστό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συναποφασίσει για την Υποσαχάρη Αφρική, την Καραϊβική, τι ε, χώρε ε, ε, ΑΚΕ και του Ειρηνικού δηλαδή. Ε, γιατί για την ώρα αποφασίζει μόνο το Συμβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να το, να το έχουμε αυτό υπόψη μας όταν θα προχωρούμε στη συζήτηση για τον προπολογισμό. Το να συμπεριλάβουμε τώρα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη στον προπολογισμό ήταν μακροχρόνιο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρούμε ότι είναι το σωστό να γίνει. Δεύτερον, θα ήθελα να επανέλθω σε κάτι που συζητήσαμε τον Απρίλιο στις Βρυξέλλες νομίζω, στρατηγικός διάλογος ε, για την ε, ε, δυνατότητα εποπτείας, εξέτασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή θέλατε μεγαλύτερη συμμετοχή στο στρατηγικό διάλογο, μπορώ να σας καθησυχάσω, να σας επιβεβαιώσω, 100% θέλουμε να συμπεριλάβουμε ε, τον, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να υπάρχει έλεγχος από το Κοινοβούλιο ε, όσο το δυνατόν γίνεται, αλλά δεν μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε στην πρόταση για νομικού λόγους. Ε, ε, ε, θέλαμε να είναι πιο στρατηγικός ο διάλογος, πιο πολιτικός και λιγότερο τεχνικός και οριοθετημένος. Θεωρήσαμε επίσης ότι θα ήταν και πιο έγκαιρο. Ο διάλογος δεν θα βασίζεται τόσο στα μέσα, αλλά στις πολιτικές προτεραιότητες εμ Χάρηκα με αυτό που άκουσα από τη Λίντα ότι θα λάβετε μία απόφαση να συνεργαστούν οι δύο επιτροπέ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπατε εκπρόσωπο, ε, οι επιτρόποι που ασχολούνται με τα εξωτερικά θέματα και οι επιτροπέ, ε, οι αρμόδιε του Κοινοβουλίου να ε, συναντηθούν όλοι μαζί. Νομίζω ότι έτσι θα έχουμε μία καλύτερη γενική εικόνα και θα έχετε κι εσεί μία συγκεκριμένη άποψη για το ρόλο σα, το ρόλο τη εποπτεία σα σε όλε τι πολιτικέ. Θεωρούμε λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να έχει μια καλύτερη εποπτεία μέσω της συμμετοχής των αρμόδιων επιτροπών του όσον αφορά του ε, τους περισσότερο τεχνικούς και τακτικούς διαλόγους. Αυτό μπορεί να γίνεται με βάση τις περιφέρειες για τη γειτονία, για την Αφρική, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Να υπάρξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όλων των μέσων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με βάση τη θεμότητα. Γιατί αν σας πω τώρα μια χώρα θα δείτε ότι υπάρχει μια πλειονότητα διαφορετικών μέσων ε, πολλών που θα πρέπει να συζητήσετε. Τρίτον, και τέλο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει ένα ε, ρόλο στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ε, τη συνεργασία μα. Θέλουμε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό. Το πλαίσιο παρακολούθηση θα ενισχυθεί από κατεξοδότηση πράξη, θα συμμετέχετε δηλαδή ε, στον καθορισμό των τομέων που πρέπει να παρακολουθούμε και θα λάβετε μάλιστα και συγκεκριμένη πρόταση. Αυτέ ήταν οι δικέ μα σκέψει, αλλά προφανώ όπω σα είπα και τον Απρίλιο, εμεί είμαστε εδώ για να ανταλλάξουμε αλλάξουμε απόψει. Εσεί προφανώ έχετε και εσεί τι σκέψει σα για το πώ μπορούμε να ενισχύσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου από εδώ και στο εξή, ε, ως το ρόλο του συνομοθέτη. Ε, αλλά ε, βεβαίως είμαστε και στη διάθεσή σας να ε, ανταλλάψουμε απόψεις για την καλύτερη συνεργασία μας στο μέλλον. Ε, να ακούσουμε και τις δικές σας προτάσεις λοιπόν ε, σε σχέση με αυτά που προσπαθήσαμε εμείς να προτείνουμε. Συγγνώμη που μακρηγόρησα. Όχι, ήταν σημαντικό γιατί εστιάσαμε πάρα πολύ ε, στα βασικά μέσα και στο βασικό υπάρχουν πολλά όμως. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Μας δώσετε και πολύ σημαντικά αριθμητικά στοιχεία και αναρωτιέμαι Είναι σημαντικό αυτό να το γνωρίζουμε για μας γιατί ε, γίνεται δημόσια συζήτηση. Και, καλό, ε, και ξέρω πάρα πολύ πο, ε, καλά πόσο σκληρά εργαστήκατε και οι δυο σας. Ντέιβιτ, θες να πεις τίποτα. Ο κύριος Νέβεν Μιμίτσα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Λίντα, αξιότιμα μέλη να εστιαστώ εν συντομία επί των αναπτυξιακών πτυχών της τομεακής προτάσεως που μας έχει υποβληθεί. Δύο στοιχεία θέλω να αναφέρω από την πρόταση. Ποιο είναι το επίκεντρο του νέου Εβραίου αυτού μέσου. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο, έχουμε σωστή ισορροπία στην πρόταση ισορροπία μεταξύ προγραμματιστέου και μη προγραμματιστέου τμήματος του εργαλείου αυτού. Η Φεντερίκα είπε ότι η ανάπτυξη πράγματι είναι στο επίκεντρο της προτάσεως του μέσου αυτού για την ε, διεθνή συνεργασία στην γειτονία. Ε, είναι ένα μέσο με παγκόσμια εμβέλεια και ταιριάζει με την φύση του νέου διεθνούς, του παγκοσμίου πλαισίου της βιώσιμης ανάπτυξης και του θεματολογίου μέχρι το 2030 και στα πλαίσια του θεματολογίου για τους ε, αναπτυξιακούς στόχους. Απομακρυνόμεθα από κάθετες απομονωμένες πολιτικές που έχουν τα δικά τους μέσα χρηματοδοτήσεως και υλοποιήσεως. Εδώ συζητούμε το θέμα της συνεκτικής πολιτικής, πολιτικής συνοχής, που ταιριάζει ε, στα μέσα της πολιτικής γειτονίας και διεθνούς συνεργασίας. Μπορείτε να δώσετε ό,τι όνομα επιθυμείτε στο νέο αυτό μέσο. Αλλά ο χαρακτήρας και η δομή του μέσου που έχει αυτό το τίτλο ε, έχει αναπτυξιακές πτυχές πάντα θα πρόκειται περί αναπτύξεως. Έχει γίνει πρόταση νομοθετική και οικονομική. Τώρα προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε την όλη δέσμη εξωτερικής δράσης και αναπτυξιακής συνεργασίας και των σχετικών παρεμβάσεων για την επόμενη επταετία. Ήδη, κατά το παρελθόν, έχουμε καθορίσει τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής. Πώς θα υλοποιηθεί αυτή η πολιτική στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συνένωσης, Συνένεσης για την Ανάπτυξη και της Παγκόσμιας Στρατηγικής. Η πολιτική είναι η ίδια, αυτή που είχαμε συμφωνήσει όλοι μας, τα κράτη-μέλη, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, μεταξύ αυτών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο. Υπάρχουν οι πολιτικές βασικό στοιχείο των αναπτυξιακών πολιτικών είναι η εξάλληψη της φτώχειας. Δεν μπορούμε να μελήσουμε το γεγονός ότι η εκρίζωση της φτώχειας παραμένει στο επίκεντρο της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Ε, είχαμε αύξηση των κονδυλίων για τα οικονομικά μας μέσα. Έχουν γίνει νομοθετικές προτάσεις για τα μέσα κανονισμός για τους κανόνες που διέπουν τις δράσεις και για τα αναπτυξιακά μας μέσα. Έχουμε μια πλήρη δέσμη μέτρων που αυτή η δέσμη ακολουθεί την αναπτυξιακή μας προσέγγιση. Στόχος είναι η ανάπτυξη και η εκρίζωση της φτώχειας. Αυτοί οι δύο στόχοι είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Αυτό το νέο ευρύτερο μέσο, κατά την άποψή μας, θα βοηθήσει και σημαντικά την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στη θέση που έχει καταλάβει που είναι ο μεγαλύτερος δωρητής για αναπτυξιακούς λόγους. Αυτό το νέο αναπτυξιακό πακέτο, το δημοσιονομικό πακέτο που εμπεριέχει πολιτικές και νομοθεσία θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε αυτό το παγκόσμιο ρόλο και να έχουμε καλύτερο αντίκτυπο σαν ε, παγκόσμιος παίκτη και στην επίτευξη των στόχων των αναπτυξιακών που έχουν τεθεί. Αυξάνοντας τις δυνατότητες εξωτερικής δράσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αναπτυξιακής συνεργασίας, συμμορφωνόμαστε με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 100 μελών να διαθέσουμε 0,7% το ΑΕΠ για την Απτυξιακή βοήθεια και 0,2% για λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Η οικονομική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ενώσεω για την επίτευξη των στόχων αυξάνεται σημαντικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των εξωτερικών δραπανών δαπανών συγγνώμη, του προπολογισμού θα εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως αναπτυξιακή βοήθεια. Θέλουμε να δίνουμε το, το ελάχιστο το 92% των αναπτυξιακών πόρων για επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Πολύ πιο φιλόδοξος αυτός ο στόχος από αυτόν που προβλέπετε τώρα. Απαντώντας λοιπόν στην ερώτηση αν χρηματοδότηση ε, αναπτυξιακή, αν θα την αποσπάσουμε και θα διαθέσουμε για άλλους μη αναπτυξιακούς στόχους, η απάντηση είναι αρνητική. Όχι. Ό,τι κάνουμε στα πλαίσια της αναπτυξιακής συνεργασίας, στο σύνολο τους οι προσπάθειες αυτές θα ενταχθούν στην αναπτυξιακή βοήθεια. Θα χαρακτηρίζεται ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. πώς θα εξευρεθεί ισορροπία μεταξύ προκατακτικού προγραμματισμού και προτάσεων ευελιξίας ούτω ώστε να υπάρχει ένα περιθώριο δράσεως σε περίπτωση απρόβλεπτων κρίσεων αυτή η ισορροπία καθορίζεται σαφώς στην πρότασή μας. Είπαμε ότι 75% τουλάχιστον των αναπτυξιακών μέσων θα πρέπει να μπορούν να, πρι, να προπρογραμματιστούν, να υπάρχει προβλεψιμότητα. Από την αρχή της περίοδου. Το υπόλοιπο αυτού του αποθέματος για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης θα εντάσσεται στην διαδικασία μέσω επιτροπολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Του ο τρόπος θα διατηρήσουμε τον πιο σημαντικό ρόλο σαν αναπτυξιακός φορέας, αλλά θα διατηρήσουμε και τη δυνατότητά μας να δρούμε ανάλογα με τις προκλήσεις που θα εμφανιστούν μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες. Η πρότασή μας καταδεικνύει σαφώς ότι η προβλεψιμότητα, η διαφάνεια, το να εστερνιστούν τα μέτρα αυτά οι χώρες εταίροι, όλες αυτές οι αρχές θα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεργασίας. Οικονομική προβλεψιμότητα θα αυξηθεί αυτή μέσω γεωγραφικού προγραμματισμού πόρων που είναι η προτιμητέα προσέγγιση για τα μέσα. Γι' αυτό προτείναμε και αυτή την προστασία ή την προσημείωση των ποσών. Έχουμε γεωγραφικούς πυλώνες, θεματικούς πυλώνες. Κινούμεθα σε ε, περιφερειακό επίπεδο, να προσημειώνονται σε περιφερειακό επίπεδο ποσά μέσω κοινού διαλόγου και μέσω διαδικασιών ελέγχου και λήψεως αποφάσεων. Και αυτό θα το κάνει το Κοινοβούλιο μέσω των διαδικασιών του προπολογισμού για τη γειτονία, υποσαχάρια περιοχή, Καραβική, Λατινική Αμερική, Ειρηνικό, Ασία. Επίσης, είχαμε καθορίσει συγκεκριμένους στόχους δαπανών. 20% των συνολικών μέσων για συνεργασία, για κοινωνική ένταξη, ισότητα των φύλων, κοινωνική ανάπτυξη, 25% για δράση για το κλίμα, 10% για μετανάστευση και μεταναστευτικές δράσεις. Αυτά είναι όλα τα στοιχεία τα οποία αποτελούν το νέο μέσο το οποίο θα μπορεί να μοχλεύει περισσότερους πόρους διαφανέστερα, με μεγαλύτερη συνοχή, με σφαιρική προσέγγιση, για να έχουν μεγαλύτερη, μεγαλύτερο αντίκτυπο οι δράσεις μας και η συνεργασία μας, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τέλος, με το νέο μέσο έχουμε πρόθεση να έχουμε περισσότερους πόρους για να διευκολύνουμε τον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο τομέα να επενδύουν μέσω απλουστευμένης αρχιτεκτονικής ε, επενδύσεων, δανειοδότησης μέσω των γεωγραφικών πυλώνων και μέχρι 60 δισεκατομμύρια μέσω ε, ταμείου εγγυήσεων ε, τα οποία, οι οποίες εγγυήσεις θα αντιμετωπίζουν τους επενδυτικούς κινδύνους που χρησιμοποιούνται για τις επενδύσεις που χρησιμοποιούνται για ε, αναπτυξιακούς στόχους. Μέσω του αποτελέσματος μόχλευσης αυτών των μηχανισμών ανάμειξης και των οικονομικών εγγύσεων θα μπορέσουμε τα δισεκατομμύρια ευρώ που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μεταφραστούν σε τρισεκατομμύρια επενδύσεων για οικονομική ανάπτυξη και βιώσιμη ε, εξέλιξη σε όλο τον κόσμο. Ε, προσβλέπω στο να ακούσω τις απόψεις σας τώρα, σήμερα, για το θέμα αυτό, αλλά και στις ε, επικείμενες διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που μαζί θα καθορίσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία πραγματικά θα καταστήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ισχυρότερο εταίρο για την αναπτυξιακή συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, για τις λεπτομέρειες αυτές κύριε Μίμητσα. Κοιτάξτε έχουμε πολλές αιτήσει από συναδέλφους να μιλήσουν. συντονιστές πρώτοι. 40 λεπτά έχουμε και λιγότερο. Οι διερμηνείς ε, στις 4.30 σχολάνε. 1,5 λεπτό έκαστος. Δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν. Και ο Ντέιβιτ έχει και σφυράκι εδώ πέρα. Λοιπόν, θα είμαστε αμήλικτοι. Παρακαλώ. Υπάρχουν συνάδελφοι που τα έχουν ξανακούσει αυτά οι συντονιστέ. Ε, το λόγο έχει ο κύριο Πρέντα, μάλλον γιατί έχει κλείσει το μικρόφωνο τη Πρόεδρου. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που έχουμε και πάλι να ανταλλάξουμε απόψει για τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα. Πιστεύω ότι φαίνεται από τις προτάσεις σας και τις ε, προτάσεις για τη νέα πολιτική γειτονία στο νέο μέσο, αλλά και το προενταξιακό το είπα, ότι ε, η κεντρική ιδέα εδώ είναι η ευελιξία. Θαυμάσια. Εδώ και καιρό στο Κοινοβούλιο ζητούμε ε, να είναι πιο ευέλικτη η χρήση αυτή των πόρων και χωρίς περιττές δυσκολίες με απλούστευση θα πρέπει να έχουμε μέσα να, δρα, να δρούμε απέναντι σε κρίσεις και διεθνείς ε, σειράξεις. Λοιπόν, από την άλλη όμως υπάρχει και το θέμα της εφαρμογής. Και υπάρχουν κάποιες ανησυχίες εδώ. Η πρώτη ανησυχία της Επιτροπής ΑΦΕΤ για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το μελλοντικό, αφορά τα όρια αυτής της ευελιξίας. Δηλαδή μέχρι πού είναι φρόνιμο και λογικό να φτάσουμε. Μήπως η ευελιξία αυτή θα καταρρύψει κάθε όριο και κάθε σύνορο. Μέχρι πού θα το τραβήξουμε. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, ε, ε, ποιος θα κάνει τη διαχείριση και το κοινοβούλιο τι ρόλο θα έχει στο νέο μέσο. Γιατί δεν αφήνει πολύ χώρο στη διαφάνεια η πρότασή σας σε ό,τι αφορά την επιλογή των προτεραιοτήτων ή ακόμα και τη χρηματοδότηση. Αυτό μας ανησυχεί. Το θέμα δεν είναι ο καθένας να τραβάει το πάπλο πάπλωμα στο μέρος του, αλλά να δούμε ε, ποιες είναι οι δράσεις και ποιοι είναι οι στόχοι. Με τρόπο διαφανή και σταματώ εδώ. Και είμαι και πολύ θλιμμένος που δεν έχω χρόνο να τα πω. Καλά. Ο Μπόγκταν Βέντα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε ε, οι δύο επίτροποι γιατί τώρα συζητούμε αυτά τα θέματα, ε, το νέο μέσο και το έργο μας και πώς θα κατανεμηθούν οι αρμοδιότητες μεταξύ ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ. Ελπίζω να καταφέρουμε να βρούμε τη σωστή προσέγγιση προς τη δική σας ε, πρόταση εγώ μιλώ από την ΔΕΒΕ. Ε, θέλουμε ένα ξεχωριστό μέσο για την ανάπτυξη και για τον έλεγχο και για την παρακολούθηση μεταξύ άλλων που είναι πάρα πολύ σημαντικά για εμάς στο Κοινοβούλιο. Αυτό μόνο ήθελα να πω. Χωριστό μέσο για την αναπτυξιακή βοήθεια. Πάρα πολύ σύντομος. Ο Νόρμπερτ Νόιζερ. Ευχαριστώ πολύ. Στα αγγλικά νομίζω ότι αυτό το ενιαίο μέσον μας δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να συντονίσουμε την πολιτική μας στις δύο επιτροπές, ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ, και να διαδραματίσουμε ένα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ίσως γνωρίζετε ότι έχουμε κάποια προβλήματα αρμοδιοτήτων, ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ, αλλά δεν είναι δικό σας γήπεδο αυτά. Ε, σίγουρα θα καταλήξουμε σε μια κοινή θέση και ένα κοινό αποτέλεσμα οι δύο επιτροπές. Άρα, έχω τις εξής δύο ερωτήσεις. Πρώτη, σύμφωνα με το άρθρο 8, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολλές αρμοδιότητες και ευρύς για τις κατεξοδότηση πράξης. Ενώ εμείς από πλευράς Κοινοβουλίου ζητούμε να υπάρχει καλύτερη και αποτελεσματικότερη συμμετοχή που να περιλαμβάνει και τη λήψη των αποφάσεων. Και το δεύτερο ερώτημα αφορά το σχέδιο, την πρόταση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, το οποίο εκδόθηκε ε, και έλεγε τα διάφορα ταμεία, αλλά από πάνω έχει μια μεγάλη σφραγίδα μετανάστευση. Τι είναι αυτό τώρα, έχετε κάνει υποχωρήσει απέναντι στα κράτη-μέλη, ότι η μετανάστευση θα καλύπτεται, ε, μάλλον θα επικαλύπτει και θα επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα. Ε, ο Τσάρλς και μετά η κυρία Σχάκε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, συγχαρητήρια στους παρόντες επιτρόπους. Τεράστια πρόκληση που αναλαμβάνουν να ενημερώσουν, εξυγχρονίσουν τα μοντέλα αυτά χρηματοδοτικά μέσα, λαμβάνοντα υπόψη τεράστιε προκλήσει μετανάστευση, αλλαγή του κλίματο, επεκτατισμό από εχθρικέ δυνάμει κλπ. που θα εμφανιστούν στο μέλλον. Και σίγουρα ε, πάντα ε, πάντα είχα μπερδευτεί με όλη αυτή την ομάδα των ε, μέσων και είμαι δύο δεκαετίε στο κοινοβούλιο. Φανταστείτε τώρα το απλό κοινό πόσο μπερδεύεται. Αυτό το λάβουμε υπόψη όσον αφορά τη διαφάνεια. Κανεί δεν τα καταλαβαίνει. Λοιπόν, απλούστευση, ενοποίηση είναι κάτι πολύ λογικό. Αλλά η ομάδα μου έχει κάποιε επιφυλάξει όσον αφορά ε, το αυτό να ενταχθεί το μέσο σε ευρύτερη αναπτυξιακή συνεργασία και ανάπτυξη. Χρειάζεται όμως ευηλιξία και καλωσορίζω την ανακοινωθήσα αλλαγή, τις σας αλλαγές που ανέφερε η κυρία Μογκερίνη, κυρίως όσον αφορά την αύξηση του προπολογισμού για την πολιτική γειτονία και προς Νότον και προς Ανατολάς και κυρίως ε, αφιερώντας πόρους προς περιφερειακή συνεργασία και υποστήριξη της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Πολύ ενδιαφέρον το παράδειγμα τη Μαυριτανία που αναφέρατε, που δείξατε ότι όπω αλλάζουν τα πράγματα, χρειάζεται ευελιξία για να κινείται κανεί γρήγορα και να μπορεί να αλλάξει τη χρηματοδότηση και τι προτεραιότητε χρηματοδοτήσεω. Ενδιαφέρθηκα ιδιαίτερα με αυτό που είπατε για ένα μέσο διευκόλυνση ειρήνη. Εγώ θεωρούσα ότι αυτή η άκαμπτη διαχώρηση μεταξύ ασφάλεια, άμυνα και ανάπτυξη, ότι υπήρχε ένα τείχο που εμπόδισε την ευελιξία. Μπορούσα να μα δώσετε παραδείγματα που θα ήταν επικοδομητικό να υπάρχει ένα μέσο εκτό προπολογισμού για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η Μαρία Τεσάκα. Ευχαριστώ πολύ. Είπατε εκπρόσωπε, κύριε Επίτροπε Μίμητσα, ευχαριστώ που ξανάρθατε. Ευχαριστούμε για την αύξηση του προπολογισμού και νομίζω ότι αυτό την χάνει ευρεία υποστηρίξεω και ευρεία εκτιμήσεω, διότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία. Παραμένει όμω το ερώτημα πώ, σύμφωνα με ποια κριτήρια τα ευέλικτα χρήματα αυτά, ευέλικτη πόλη θα χρησιμοποιούνται. Ποια θα είναι η εφετηρία, ξεσπάει μια κρίση. Πότε αποφασίζουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το Ταμείο Ευελιξία και πώ αποφεύγουμε να αδειάσει το Ταμείο μετά από δύο χρόνια κρίσεων όταν έχουμε ένα κύκλο προπολογισμού 7 ετή. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό για μένα. Αυτό που δεν θέλαμε να δούμε εδώ στο Κοινοβούλιο είναι επανάληψη των πρακτικών τη συμφωνία με την Τουρκία ή την εμφάνιση καταπιστευμάτων όπου τεράστιοι πόροι ε, χρησιμοποιούνται χωρί καμία υποπτία από τη δική μα πλευρά. Οπότε ε, είναι πολύ καλό το ότι οι αναπτυξιακοί πόροι βρίσκονται υπό κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά δεν απάντησε κάθε ερώτημα όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Θα πρέπει επίση να κατανοήσουμε ότι λόγω των περιορισμών των επτατών κύκλων του προπολογισμού είμαστε περιορισμένοι όσον αφορά τι αποφάσει σχετικά με το τι θα θέσουμε στου ανθρώπου για το 2026, στους αρμόδιου, Παραδείγματο χάρη. Επαναλαμβάνω, πρώτερε προειδοποίησει. Υπάρχει κίνδυνο ότι θα γίνει πολιτικός, η πολιτική καθοδήγηση, θα γίνει η λαϊκιστική καθοδήγηση, θα καθοδηγείται από βραχυπρόθεσμα συμφέροντα και μακροπρόθεσμα και τους συσχετισμούς θα τους χάσουμε, τις διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων θεμάτων και οριζόντια ζητήματα θα χάσουμε, ε, δεν θα έχουμε πλέον τον έλεγχο. Δεν είδαμε κάποια κατεξουσιοδότηση πράξη, στρατηγική διάλογη, δεν υπήρξαν επιτυχείς ε, κατά γενική ομολογία. Θα πρέπει να επεξεργαζόμεθα κύκλους που γνωρίζουμε. Συγγνώμη, τελειώνω ε, οποιαδήποτε έκθεση για διεύρυνση για ανθρώπινα δικαιώματα, συστάσεις από παρατηρητές εκλογών να λαμβάνονται υπόψη, ούτω ώστε να ταιριάζουμε την πρωτοβουλία που θα πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του φυσικού κύκλου που υφίστανται, με κοινοβουλευτικό έλεγχο και ε, χειρισμό. Ευχαριστώ. Ο κ. Γκέρενς, πολύ καλά συνοψιστήκαν όλα. Τι πρέπει να γίνουν στα πλαίσια των δύο επιτροπών. Δεν θα αναφερθώ στο θέμα αυτό. Ε, είναι πολύ είναι πολιτικό το θέμα. Πιστεύω ότι ο πραγματικός που μας εμποδίζει και είμαστε σε, κύκλο είναι το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη και βρισκόμαστε σε φαύλο κύκλο. Όταν θέλουμε να καθορίσουμε μετά το κοτονού την εντολή είναι μια χώρα ε, που θέτει τροχοπέδι. Είναι υπεριαλισμό αυτός και καταστρέφει την Ευρώπη μας Θα ενισχύσουμε λοιπόν το ρόλο των κρατών μελών ε, όσον αφορά την λειτουργία αυτή της ε, των προσπαθειών. Λοιπόν, αναλαμβάνονται ε, ε, δεσμεύσεις που δεν τηρούνται και όταν ζητούμε με τα κράτη να δικαιολογήσουν γιατί τελικά ε, βγαίνουν εκτός ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρνούνται ακόμα ε, αν υποτίθεται κάτι τέτοιο αναφέρεται στις συνθήκες. Και αυτό που χάνει σε αυτέ τι περιπτώσει τελικά είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ηττημένο. Δεν ξέρω αν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη θα συμπεριληφθεί. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Έχω αμφιβολίε, ελπίζω ότι θα, ληφθεί, θα συμπεριληφθεί. Αν δεν συμπεριληφθεί, θα συνεχίσουν τα πράγματα όπως τώρα, τα κράτη-μέλη θα αποφασίζουν αυτό που θα μπορεί να πληρώνει τα Ευρωπαϊκά, Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Ταμείο Ανάπτυξης. Λοιπόν, αν ενταχθούν τα πάντα, θα κάνουν τα πάντα για να μην υπάρχει καμία κατεξοδόση πράξη, ούτω ώστε και εκεί να μπορέσουν να, θέσουν, να παίξουν το ρόλο του στου Αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί το λέω αυτό, Διότι θα ήθελε η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βλέπουν το βασικό του σύμμαχο στο Κοινοβούλιο. Έχουμε συμφέρον να είμαστε σύμμαχοι και έχουμε συμφέρον επίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει μέχρι πού θα προχωρήσουν αφορά την ευελιξία. Αυτό αναφέρθηκε από του προλαλήσαντε αγορητέ. Η ερώτησή μου είναι απλή. Όταν η ευελιξία μπαίνει σε ανταγωνισμό με τα προνόμια τα κοινοβουλευτικά, τι θα, σε τι θα θέσετε προτεραιότητα σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για να απεμπλακεί αυτή η κατάσταση άπαξ διαπαντό. Διότι είναι η κορονίδα τη εξωτερική μα πολιτική και τα κράτη-μέλη τα οποία μέχρι τώρα διαχειρίζονται 80% του ε, δημοσίου χρέους το αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, θέλουν τα πάντα να διαχειριστούν με μία μέθοδο ε, που δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Οι πράσινοι, οι συντονιστές έφυγαν. Είσαι στον κατάλογο. Και σκοράω. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ εκ νέου τους Επιτρόπους Έχετε γίνει Φάμπιο Καστάλτο. Δεν είμαι ο Καστάλτο, δεν είμαι ο Καστάλτο. Δεν πειράζει, είναι καλός φίλος. Κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ την Επίτροπο, τους Επιτρόπους που είναι εδώ και επαναλαμβάνω αυτό που ήδη είχα επαναλάβει και είχα αναφέρει την προηγούμενη φορά σαν αφορά ε, το προβλήματα όσον αφορά την ευελιξία. Συμφωνώ αυτά που είπε ο κύριο Σάλ Γκροέντ, όσον αφορά το πρόβλημα ευελιξία με κοινοβουλευτικό έλεγχο. Από την άποψη την κοινοβουλευτική είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε με ποιο τρόπο κατευθύνονται αυτοί οι πόροι και να μπορούμε να ελέγχουμε ε, τις διάφορες κατανομές των ποσών και να βλέπουμε πώς δαπανώνται. Λοιπόν, αν και εξηγήσει σας ε, είναι απόλυτα αποδεκτές, εγώ πιστεύω που κοινοβουλευτική άποψη υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα μετά που αφορά τους πόρους. Ε, θα, λοιπόν, μιλάτε για μια αύξηση των ε, πόρων. Θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα από πού φτάνουν αυτοί οι πόροι. Από το Ταμείο της Ανάπτυξης και θα μετατεθούν στο ενιαίο μέσο ή προβλέπονται και μεγαλύτερες εισφορές από πλευράς κρατών μελών. Διότι αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι σαφέστατο. Αυτό το Ταμείο για τις κατεπίγουσες ανάγκες, από πού θα τροφοδοτείτε θα ήθελα κάποια διευκρίνηση μεγαλύτερη ε, όσον αφορά την προέλευση και χρήση των πόρων. Όσον αφορά την ευελιξία, επιβεβαιώνω αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως. Ευχαριστώ. Now we've had about 11 Ακούσαμε περίπου 11 ε, παρεμβάσεις και έχουμε άλλες 12. Μήπως μπορείτε να είστε κι εσείς σύντομοι, θέλετε να απαντήσετε τις πρώτες. Α, θα τι απαντήσετε όλες μαζί. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να σας παραφορτώσω με το να κρατάτε σημειώσει. Συνεχίζουμε τότε. Δεν μπορώ να το χωρίσω σε ομάδες. Θα τα πάρουμε τη σειρά προτεραιότητα. Ο Αρνελίτς, ευχαριστώ πολύ για την ανταλλαγή αυτή απόψεων. Πάρα πολύ σύντομο θα είμαι. Μια ερώτηση έχω. Συζητήσαμε πάρα πολύ το ICSP αυτό είναι ένα μέσο που θέλουμε το έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά τι γίνεται, γιατί η χρηματοδότηση είναι διαφορετική, γιατί δεν υπάρχει πια το DCI, πώς θα μοιράσουμε τις αρμοδιότητες και από το Κοινοβούλιο Α, ξέρετε ότι υπάρχει μια γερμανική πρωτοβουλία διτή ε, από, την, από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Υπουργείο Εθνική Αμήνη. Να ρωτήσουμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη και πώ ε, χρηματοδοτούν αυτή τη βοήθεια. Σα ευχαριστώ που μιλήσατε και για το κλίμα. Ε, πριν από λίγες μέρες ήταν εξαιρετική αυτή η διάσκεψη για το κλίμα και χτες είχαμε και την έκθεση για την κλιματική διπλωματία στο Κοινοβούλιο. Τώρα θα πρέπει να ενταθεί ο διάλογος και για τη χρηματοδότηση ζητούμε ε, ε, να αναλαμβάνουν ε, αυτό το έργο οι κατατόπου αντιπροσωπείες μας που έχουν και το προσωπικό και τις δυνατότητες και μπορούν να συνεργάζονται με τις πρεσβείες. Δηλαδή να μην γίνονται όλα αυτά σε επίπεδο κυβερνήσεων αλλά σε τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι και τα δημαρχία. Μπορείτε να το βάλετε αυτό στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο γιατί και εμείς ως κοινοβούλιο έχουμε τις σχέσεις μας με τις αντιπροσωπείες και θα πρέπει να δούμε πώς θα ε, γίνουν αυτά και πώς θα ε, χωριστούν οι αρμοδιότητες. Ευχαριστώ κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ δύο συντονιστές ε, αντικαθιστώ που δεν μπορούν να είναι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ακούσουμε αυτό που είπατε, είπατε εκπρόσωπε σε σχέση με τους στόχους και τις ανάγκες και μετά αποφασίζεται το μέσο. Όμως εδώ έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις, σημαντικές ερωτήσεις. Θα δουλέψει πράγματι έτσι το σύστημα. Άκουσα μία πάρα πολύ σαφή παρουσία... Ε, για το κέντρο ανάπτυξης, ε, πολιτικής ανάπτυξης. Ε, θα ήθελα λοιπόν όλα αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα ε, που προσπαθείτε να τα δείτε και μέσα από το πολιτικό πρίσμα θα αντιμετωπιστούν. Εμένα μου φαίνεται πραγματικά το περίεργο το ότι κάποιες πολιτικές προτεραιότητες ε, συγχωνεύονται με γεωγραφικά θέματα το θεματικό πρόγραμμα και οι παγκόσμιες προκλήσεις είναι τρία δις, ενώ τα γεωγραφικά ε, προγράμματα δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια ε, αντιπροσωπεύουν. Πώς θα εξασφαλίσουμε και σε αυτή την περίπτωση ότι οι θεματικές προτεραιότητες θα επιφέρουν μια αλλαγή στο πλαίσιο της, ε, των στόχων αηφόρου ανάπτυξη, όπως είπε και ο κύριος Μίμητσα. Μιλήσατε για τους στόχους αυτούς και είπατε ότι θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ε, εντάξει, αλλά για ποιο λόγο στην πρόταση, τουλάχιστον εγώ, δεν είδα τίποτε που να αφορά τους ε, στόχους αηφόρου ανάπτυξης. Ε, δεν αναφέρεται εξ όσων κατάλαβα ο στόχο, Ευχαριστώ Χάιντι. Η κυρία Ζόφκο. Thank you. Thank Ευχαριστώ πολύ να συνεχίσω το ερώτημα αυτό ε, προς τον Επίτροπο Μίμητσα να μας εξηγήσει μαζί με την ε, ύπατη εκπρόσωπο Μογκερή να μας πει ποια είναι ο συντονισμός επιτόπου αυτών των στόχων ε, αηφόρου ανάπτυξης μεταξύ των διαφόρων φορέων πόσα χρήματα και πόσα μέσα εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσεων, μέσων να συμπεριλαμβάνετε στις ε, ε, συνεργασία σας ε, με το εξωτερικό γιατί υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις και το θέμα της ασφάλειας και της ειρήνης. Ποια γίνεται λοιπόν, πώς γίνεται ο συντονισμός με τις πρεσβείες των άλλων χωρών και πόσα χρήματα επενδύονται στο προσωπικό και στους διπλωμάτες που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα μέσα για τα οποία μιλούμε. Ο κύριος Κορνιέ. Ευχαριστώ προτείνετε συγχώνευση σε ένα ενιαίο μέσο. Πιστεύετε ότι έχετε επαρκέ προσωπικό τόσο σχηδές για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλη αυτή τη διαφοροποίηση των προγραμμάτων σε τέτοιε γεωγραφικέ περιφέρειες. Νομίζετε ότι αυτό είναι καλό. Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη, ε, θα έπρεπε να χρηματοδοτείται από τον Γενικό Προϋποτολογισμό. Ε, ε δηλαδή, συνεισφορά των κρατών μελών, ε, πώς θα γίνει γίνει όμως αυτό, θα συνεχίσουν ε, να συνεισφέρουν για το ίδιο ποσοστό ή θα υπάρχει μία μείωση ε, του συνολικού αναπτυξιακού προπολογισμού, γιατί θα γίνεται κάποια χρηματοδότηση των ίδιων στόχων από αλλού. Τρίτη ερώτηση. Είπαμε ότι, ο, είναι βασική η αναπτυξιακή χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις τρίτες χώρες, όμως αν δείτε στην πράξη τα νούμερα, είναι διαφορετικά από τα νούμερα που μας είπατε εσείς. Πολλές χώρες εταίροι δεν έχουν τη δυνατότητα της διαχείρισης της οικονομικής για να ανταποκριθούν στις, ε, δικής μας, ε, στις δικές μας απαιτήσει. Χρειάζεται λοιπόν και κατάρτιση και εκπαίδευση να υπάρξει υπάρξει δηλαδή, να υπάρξουν σεμινάρια, ε, να υπάρξουν σεμινάρια ε, βασικής εκπαίδευσης και των τοπικών αυτοδιοικήσεων των κρατών ε, που είναι δικαιούχοι για να μπορέσουν να ζητήσουν τα χρήματα που εμείς θα τους δώσουμε και να μπορέσουμε να επιτύχουμε τα νούμερα που μας αναφέρατε. Ευχαριστώ πολύ. Άννα Γκόμες. My, my are... Οι ανησυχίε μου αφορούν τη στρατηγική κατεύθυνση η εκπρόσωπο εκπρόσωπος πρέπει να δώσει μια στατική κατεύθυνση και να ενταχθεί στην προσέγγιση. Για όλες τις δομές. Αυτό δεν αφορά μόνο θέματα ανάπτυξης και εξωτερικής δράσης, αλλά και άλλους τομείς. Εμπόριο, θέματα εσωτερικών πολιτικών ελευθεριών. Δεν θέλουμε βραχυπρόθεσμη θεώρηση που είναι αντιπαραγωγική παράνομη δράση για μετανάστευση. Αυτοί που συζητούν τα κράτη-μέλη. Πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επανάληψη των φοβερών συμφωνιών όπως με την Τουρκία. Χρειαζόμαστε αυτή την κατεύθυνση που πρέπει να προέλθει από την ύπατη εκπρόσωπο. Θα σας στηρίξουμε σε κάτι τέτοιο. Οποιαδήποτε στρατηγική για τους στόχους της σχετίας θα αφορούν σωστή διακυβέρνηση, κοινωνία των πολιτών, δημιουργία δυνατοτήτων για εκείνους που πρέπει να κάνουν τις, χω... τις κυβερνήσεις να λογοδοτήσουν για διαφθορά, ανθρώπινα δικαιώματα, χρηστή διακυβέρνηση κλπ. Δεν αφορά τις ανοησίες που είχαν αρνητικά αποτελέσματα και που γι' αυτό το λόγο προσπαθεί ο κόσμος να ξεφύγει από την Αφρική και από αλλού. Τέλος, πρέπει να υπάρχει έλεγχο για, για το μέσο για την ειρήνη στην Αφρική. Πώς θα γίνει όμως αν είναι εκτός προπολογισμού τα χρήματα. Ευχαριστώ. Μπορούμε να μάθουμε το ETF. Ερίκε Γκερέρο. Ευχαριστώ, ναι. Από τότε που αρχίσαμε αυτή τη συζήτηση, επικεντρωθήκαμε στα μέσα αποκλειστικά. Και αυτό είναι λάθος εστίαση, πιστεύω τελικά τα μέσα είναι ακριβώς επιχειρησιακά μέσα για να φτάσουμε στους στόχους μας που είναι οι πολιτικές και θα πρέπει να συζητήσουμε ακόμα πολλά για το ποιο ρόλο διαδραματίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι παγκόσμιος ε, πρωταγωνιστής η αναπτυξιακή βοήθεια. Έχει αλλάξει πάρα πολύ ο κόσμος από τότε που εγκρίναμε τις προηγούμενες ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Προχωρήσαμε στην εξωτερική πολιτική, αμυντική πολιτική, πολιτική ασφαλείας αλλά η αναπτυξιακή πολιτική εκεί παραμένει μια, ε, μια ήπια δύναμη που θέλει η Ευρώπη να συνεισφέρει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στον κόσμο. Αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε ακόμα πολύ την πολιτική ταυτότητα της αναπτυξιακής πολιτικής που είναι και στην συνένεση για την ανάπτυξη και στις συνθήκες αλλά και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Και τα δύο θα πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή να ενισχύσουμε το ρόλο της ανάπτυξης στην ε, παγκόσμια πολιτική της Ένωσης αλλά να ενισχύσουμε και την ταυτότητά της και να τη διαφυλάξουμε αυτής της πολιτικής ανάπτυξης βάσει των ίδιων των αρχών και ε, στόχων της. Αυτό πώς γίνεται με τη διατήρηση της χρηματοδότησης, με μακροπρόθεσμους στόχους, αλλά και υπερασπίζοντας ε, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτό είναι που θα πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Τώρα το αποτέλεσμα αν θα είναι ένα το μέσο ή πολλά θα είναι ε, η κατάληξη αυτής της δουλειάς και όχι αφετηρία απριόρι. Ο κύριος Σοσιένιτς. Ε, Ευχαριστώ. Εμεί στην Πολωνία πολύ συχνά λέμε ότι Μπορεί κάποιος να είναι πολύ γενναιόδωρος εις βάρος σε άλλον. Και νομίζω ότι εδώ έτσι συμπεριφερόμεθα. Θέλετε να δαπανίσετε τα χρήματα του φορολογούμενου σε όλο τον κόσμο χωρίς να πετυχαίνετε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και τον περισσότερο χρόνο οι φορολογούμενοι δεν έχουν την παραμικρή ιδέα τι τρέχει εδώ πέρα. Νομίζω ότι δεν έχετε δικαίωμα να το κάνετε αυτό. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει ένα δημοψήφισμα για να ξέρουμε αν οι φορολογούμενοι συμφωνούν να εργάζονται για να χρηματοδοτούν τις κυβερνήσεις που είναι διεφθαρμένες των τρίτων χωρών. Δεν πιστεύω ότι συμφωνούν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Και εσείς οι ίδιοι, επανειλημμένα σε διάφορες εκθέσεις, ομολογείτε ότι τα χρήματα αποτέλεσαν αντικείμενο κακής διαχείρισης. Κάποιες χώρες πήραν πολλά χρήματα, Φερρυπίν δεν έκαναν τίποτα με αυτά τα χρήματα. Προφανώς μπορούμε να επενδύσουμε περισσότερα στην αλλοδαπή, αλλά όλα αυτά θα έπρεπε να δίνουν αποτελέσματα, συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα πρέπει να έχουμε επιχειρηματική λογική που ακολουθούμε. Εδώ όλα αυτά που λέμε είναι παράλογα. Δεν έχουν την παραμικρή λογική. Εν ονόματι τίνο να γίνουν όλα αυτά. Εν ονόματι κάποιων αυθαίρετων κριτηρίων που έχετε φανταστεί. Ε, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε ο τρόπο να δαπανείτε τα χρήματα, δαπανάτε τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων ε, εκτό των συνόρων όταν έχουμε προβλήματα σημαντικά εδώ πέρα. Ελπίζω να μην εφαρμοστεί τελικά αυτή η πολιτική. Ευχαριστώ. Έλλη Σλάιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκτιμώ τις προσπάθειες που γίνονται για απλούστευση του πλαισίου, που είναι αρκετά περίπλοκο. Συμφωνώ όμω με τι ανησυχίε των άλλων συναδέλφων, εξαρτάται πώ θα γίνει αυτό. Είπατε εκπρόσωπο αναφέρθηκε στι τάσει τι οποίε είδαμε τελευταία χρόνια και συζητήσαμε επινειλημμένα και με τον Επίτροπο Μίμητσα Δηλαδή οι αναπτυξιακέ δαπάνε να μετακινούνται προ βραχυπρόθεσμου στόχου ε, στα κάτι μελη Να σταματήσει η μετανάστευση, να γίνεται καλύτερη διαχείριση των συνόρων, Φερρυπίν, που δεν ταιριάζει με την εκρίζωση τη φτώχεια. Φοβούμε ότι σε ένα μεγαλύτερο κουρβανά μαζί με άλλε πολιτικέ τα συμφέροντα τα εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα επικρατήσουν των αναπτυξιακών στόχων. Και είναι απογοητευτικό που τα κράτη-μέλη δεν θέτουν αρκετά χρήματα και όχι μόνο αυτό, αλλά ασκούν και πιέσει να παίρνουμε την ψυχική βοήθεια και να την αφιερώνουμε για την ασφάλειά τους. Δεν μπορούμε να την θεσμοθετήσουμε αυτή την τάση και ανησυχούμε για την έλλειψη σαφήνειας για τα κριτήρια για την κατανομή των πόρων και για το δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου και με το καταπίστευμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται πραγματικά επί τόπου. Υπάρχουν πραγματικά προγράμματα αναπτύξη όπω στην Ουγγάντα που για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά και προγράμματα όπω στη Λιβύη και στον Ήγηρα που έχουν άλλο προσανατολισμό και είναι σαφέ και δεν θα πρέπει να πληρωθούμε αυτά τα χρήματα. Και οι στόχοι τη χιλιετία θα πρέπει να είναι ένα γενικότερο πλαίσιο που θα καθορίζει την πορεία των μέσων, αλλά αυτό αναφέρεται μόνο ακροθυγώ και δεν θεωρείται σαν βασικό πλαίσιο για υλοποίηση και έλεγχο. Τι είδου μέτρα διαφύλαξη προβλέπετε, τόσο ώστε αυτό να είναι περισσότερη ευκαιρία παρότι κίνδυνο. Για μένα, όπω τα βλέπω τα πράγματα, είναι περισσότερο κίνδυνο. Ο κ. Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο πράγματα. Πρώτον, είμαι μεταξύ εκείνων που είμαστε ικανοποιημένοι γιατί έχουμε πόρους που μπορούν να βοηθήσουν ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση για την οικονομία, το εμπόριο, τη βιομηχανία και αυτό δεν ήταν καθόλου αυτονόητο γιατί είναι και ισχνή οι πόροι που έχουμε. Δεύτερο, στο Κοινοβούλιο υπάρχουν δύο σκολές σκέψεις. Ε, ορισμένοι είναι υπέρ των πολλών μέσων ε, και εγώ είμαι μέλος αυτής τη Επιτροπής που είναι και αντιπαθητική, της Επιτροπής Ελέγχου των Προπολογισμών που θεωρούν ότι χρειάζεται εξορθολογισμός. Το έχει πει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο. Ο κύριος Γκερέρο πολύ ωραία το υπογράμμισε. Έχουμε, ε, τις, οι πολιτικές είναι στην υπηρεσία των μέσων ή τα μέσα τα χρηματοδοτικά στην υπηρεσία των διαφόρων ε, πολιτικών ανάπτυξης. Το δεύτερο προφανώς και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στην εκπόνηση αυτών των χρηματοδοτικών μέσων. Ε, η κυρία Μογκερίνη με πολύ χάρη μας είπε πώς θα σκεφτούμε να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο. Κυρία Μογκερίνη, ξέρουμε τι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να δίνουμε απλώς την ευλογία μας και σε σημαντικά ποσά και μετά βάσει της αρχής της ευελιξίας με την οποία συμφωνώ να μείνουμε εκτός νυμφώνος. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει ένα χώρο και έχει ένα χώρο και τα διευρεμένα μας προεδρία των δύο επιτροπών θα ορίσουν εισηγητέ. Θα πρέπει λοιπόν να προβληματιστούμε, να σκεφτούμε τι θέλουμε και η Κομισιόν που έχει δικαίωμα πρωτοβουλία να κάνει τις προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ειρήνα Γκίλ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία, πιο ευελικτά μέσα, ούτω ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε νέε προκλήσει. Η παρούσα πρακτική που ακολουθούμε όσον αφορά στρατηγικό διάλογο και προγραμματισμό δύο φορέ το χρόνο επί επταετία και πρόσβαση σε επιτροπολογία είναι κάτι που είναι ανεπαρκέ. Θα έλεγα λοιπόν ότι καλωσορίζω αυτά που μα είπατε, τι διαβεβαιώσει που δώσατε, είπατε εκπρόσωπε, ότι θα έχει μεγαλύτερο έλεγχο το Κοινοβουλίο στον αφορά τι προτάσει. Δεν είναι ξεκάθαρο για μένα το εξή. Στη διαδικασία λήψη αποφάσεων, πότε μπορούμε να παρέμβουμε στα διάφορα, στις διάφορες διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ή πώς θα λειτουργήσει αυτό στο μέλλον. Διότι αυτό θα αλλάξει το ρόλο κάπως. Θα πρέπει να ξέρουμε τι αντίκτυπο θα έχει. Ε, δεν πιστεύω ότι έχω καταλάβει καλά το πώς οι πόροι για συγκεκριμένους στόχους θα διαφυλάσσονται και συμμερίζομαι πολλές ανησυχίες που εξέθεσαν συνάδελφοι. Δηλαδή, είναι πραγματικά σημαντικό η ευελιξία να είναι εσωτερική και δεν θα μειώνει ε, το γενικό κουρβανά ανεξάρτητα από τις που θα αντιμετωπίζουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να έχουμε ευελιξία για νέα προβλήματα και νέε προκλήσει, Παρακαλώ όμω να μην παίρνε, αφαιρείτε τι πολιτικέ προτεραιότητε για τη γειτονία, Λατινική Αμερική, Ασία ή για οποιαδήποτε άλλη προτεραιότητα. Είναι σημαντικό αυτό να αναθεωρούμε και να προσαρμοζόμεθα, αλλά να μην αφαιρείται ποσά. Επίσης να πω ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ διαφόρων πολιτικών προτεραιοτήτων. Και αυτό καμιά φορά λείπει. Και ορατό της. Σας παροτρύνω, κοιτάξτε το αυτό, διότι συχνά βλέπουμε προγράμματα, τα εξετάζουμε και είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε εάν έχει υπάρξει σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά. Και θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πραγματικά σημαντικό αυτό για μας, για τις πολιτικές προτεραιότητες, να είμαστε θεμελιώδους σημασία στην ε, εφαρμογή της ευελιξίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Νίνα. Ο κύριος Φουντουλίκα. Φρουντουλίκα. Φρουντζούλικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Υπόθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερο δωρητή ε, σε όλο τον κόσμο για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια. Παράλληλα όμω βλέπουμε την ε, υποβάθμιση του περιβάλλοντο, ότι δεν υπάρχουν πλέον αρκετοί πόροι σε πολλά μέρη στον κόσμο. καταναλώνονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια μέχρι το, τον Αύγουστο και μετά είμαστε επιπιστώσει μέχρι το τέλο τέλος της χρονιάς. Ε, θα ήθελα λοιπόν να κάνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περίπτωση ετήσιου ενδεικτικού προγράμματος ε, εθνικού ε, ενδεχομένως να πρέπει να μπορούμε να εφαρμόζουμε όλες τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίες και με τρίτες για την εφαρμογή και την προώθηση των στόχων αηφόρου ανάπτυξης. Είναι σημαντικό και τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν ε, τους στόχους ε, ανάπτυξη, ανάπτυξης, γιατί υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν τους ε, σέβονται. Παράλληλα, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή και η Ευρωπαϊκή Ένωση, Εμεί όλοι από κοινού πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, η αύξηση του πληθυσμού της Αφρικής, και το λέω αυτό σε σχέση με τη μετανάστευση, από 1 δις 288 εκατομμύρια το 2018 μέχρι το 2025 ο πληθυσμός θα αυξηθεί κατά 200 έως 500 εκατομμύρια άτομα. Άρα χρειαζόμαστε μια στρατηγική προσέγγιση για το ζήτημα αυτό που θα, ενημερώσει, θα επηρεάσει πάρα πολύ το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βάιταλ. Ε, ευχαριστώ. Κυρία Μογκερίνη, ήσασταν αρκετά επιτυχής ε, κατά τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες ε, στη διαμεσολάβηση σε διάφορα μέρη όπως το το Ιράν και στη Μακεδονία, στην Ελλάδα και σε άλλα προβλήματα τα οποία προσπαθήσατε να διαμεσολαβήσετε. Έχω όμως ε, την αίσθηση ότι αυτό που ε, χρειαζόμαστε ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής μας θα ήταν μία μόνιμη ομάδα συμφιλίωσης, μία για διαμεσολάβηση και μία για τη διαμόρφωση στρατηγικής ε, και την ανάληψη πρακτικών μέτρων ε, για τις παγιωμένες ε, συγκρούσεις στη γειτονιά μας. Δεν είναι μόνο δηλαδή η καθημερινή συμμετοχή δική σας προσωπικά και της δική της ομάδα, σας ομάδας. Θα χρειαζόμασταν ανθρώπους που θα αφιερωθούν σε μια μακροπρόθεσμη, μακροχρόνια δουλειά για το θέμα αυτό. Ο κύριος Φρόντ, Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Προσπαθώ ακόμα να συγκεντρώσω όσο γίνεται περισσότερες ψήφους για την έκθεσή μου για τα Ηνωμένα Έθνη αύριο. Ε, και αυτό μου πήρε λίγο περισσότερο χρόνο από όσο υπολόγιζα. Δεύτερον, καμιά φορά όταν συμμετέχω σε τέτοιες συνεδριάσεις τα βλέπω υπό την ιδιότητα του δημοσιογράφου που ήταν η προηγούμενη δουλειά και λέω Θεέ μου πιστεύουμε πραγματικά ότι τον νοιάζει τον κόσμο ποιος έχει αναλάβει ένα συγκεκριμένο έργο και ποιος το εκτελεί. Αυτό που τους νοιάζει είναι τι γίνεται και τι κάνουν για μας. Το είπα και χτες. Στον καγκελάριο Κούρτς που έκανε την παρουσίασή του στην Ολομέλεια. Τον καγκελάριό μας. Και του είπα το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε εκτός από αυτή την πολιτική της κινδυνολογίας ε, που φαίνεται ότι τους έχει γίνει η ιδέα στα πολιτικά κόμματα, γιατί να μην αρχίσετε να εκπονείτε ένα σχέδιο Μάρσαλ για την Αφρική. Για την Αφρική, με την Αφρική, εν πάση περιπτώσει, στην Αφρική. Αυτό θα σας δώσει πολύ περισσότερη αξιοπιστία και κύρος στον κόσμο, αντί να κάνεις αυτά που κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, ε, Έχω ενθουσιαστεί και με έχει συναρπάσει μια έκθεση που είδα πρόσφατα για φωτοβολταϊκά και λύσεις εκτός ε, συνδεδεμένου δικτύου στην Αφρική, off-grid. Αμερικανικές εταιρείες, μικρές εταιρείες, μικρομεσαίες εταιρείες. Microcredit. Βοηθάνε το λαό εκεί με μικροπιστώσεις, με ε, συσσωρευτές, μπαταρίες για να μπορούν να έχουν ε, αντλίες ε, για νερό, που να δουλεύουν όλη τη μέρα, φυσικά όχι τη νύχτα, ε, και έχουν και νερό για την άρδευση αλλά και για την ίδρυυση. Και μπορούν να παράγουν τρόφιμα. Οπότε δεν χρειάζεται να φύγουν από εκεί για να έρθουν εδώ. Εμείς γιατί δεν τα κάνουμε αυτά. Εμένα ένα σχέδιο, σχέδιο Marshall. Thank you. Thank you, I think we probably do. Ευχαριστώ, και Μάλλον θα το κάνουμε. Το κάνουμε κι εμείς, γιατί έχω δει και εγώ τέτοια δικά μας project. Φεντερίκα. Thank you. I'll try to be brief. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και θα αφήσω στον Εύεν ε, τις, ε, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με την ανάπτυξη. Καταρχάς, οι πολιτικές ε, προτεραιότητες ε, είναι σαφώς, ε, έχουν αναφερθεί σαφώς στην πρόταση. Τώρα να δούμε κατά πόσο θα δούμε αν θα υπάρξουν άλλες εξελίξεις, αλλά είναι πολύ σαφείς οι προτάσεις μας και για τις πολιτικές προτεραιότητες και για τα χρήματα που θα δοθούν σε αυτές τις προτεραιότητες. Θα δώσω ένα άλλο παράδειγμα για το λόγο για τον οποίο θα ήμουν ε, υπέρ ενό ενοποιημένου και απλοποιημένου μέσου, αλλά και του κοινού προγραμματισμού με τα κράτη-μέλη. Όλοι μιλούν για ένα σχέδιο Marshall για την Αφρική. Μπορώ να σας ρωτήσω, έχετε καμία ιδέα πόσα χρήματα επενδύουμε στην Αφρική με όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού, συν τα κράτη-μέλη, 20 δις ευρώ κατέτος. Αυτό δεν είναι σχέδιο Μάρσαλ είναι ένα σχέδιο μας, αλλά το βλέπουμε μέσω κατακαιρματισμένων ε, φακών. Δεν βλέπουμε δηλαδή το πλήρες φάσμα των όσων κάνουμε, ούτε οι εταίροι μα, γιατί προέρχεται από χίλια, διαφορετικέ διαφορετικές ε, ε, διόδους. Ε, αν λοιπόν υπάρχει κατακαιρματισμό και ο αντίκτυπο είναι πολύ μικρότερος. Δεν είναι μόνο η Μαυριτανία, είναι ο πολιτικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει κανεί με την επένδυση που ούτω ή άλλω κάνει. Ε, μέσω των πολιτικών προτεραιοτήτων. Όσον αφορά τα καταπιστεύματα, συμφωνώ απολύτω. Ένα από του λόγου για του οποίου προτείναμε αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση και αυτή την απλοποίηση είναι για να αποφύγουμε ότι στο μέλλον θα πρέπει να εφεύρουμε μέσα τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί πριν από 7 χρόνια. Και αυτό είναι ε, ένα από τους λόγους ε, της συγχώνευσης κάτι, κάτι ακόμη για συγκεκριμένες ερωτήσεις για τη μετανάστευση αν πρόκειται να επισκιάσει τα πάντα. Όχι στην πρόταση. Σίγουρα όχι στην πρόταση. Τώρα το πώς θα προκύψει, πώς θα, προκύψει αυτή η πρόταση στο πλαίσιο της διαδικασίας ε, λήψη αποφάσεων που έχουμε ενώπιόν μας εξαρτάται και από τα κράτη-μέλη. Να δούμε τι θα γίνει. Αλλά είμαι υπέρ του να διατηρηθεί η μετανάστευση, η εξωτερική δράση για τη μετανάστευση όσο ε, τμήμα τμήμα των εξωτερικών μας δράσεων με ένα συγκεκριμένο ποσό αφιερωμένο σε αυτή 10% που είναι αύξηση ε, του ποσού που επενδύουμε τώρα, αλλά και μια ενσωματωμένη προσέγγιση μαζί με την ανάπτυξη, γιατί διαφορετικά γνωρίζουμε ότι αυτά τα χρήματα υπάρχει ο κίνδυνος να μην πάει ε, το, τα, να τα χρήματα αυτά ε, στη σχέση μεταξύ των αιτίων της μετανάστευσης και της ανάπτυξης. Γι' αυτό χρειάζεται επένδυση. Δεν είναι επένδυση στη διαχείριση της μετανάστευσης που λύνει τα προβλήματα της ανάπτυξης. Αντιστρόφως, το να επενδύσουμε στην, στην, ε, στην ανάπτυξη μας βοηθάει βοηθά στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Όσον αφορά την, την διευκόλυνση για την ειρήνη. Ε, είπατε ότι είπαμε ότι θα είναι εκτός προϋπολογισμού, μου ζητήσατε παραδείγματα κατά τη γνώμη μας ε, θα αντικαταστήσει το μηχανισμό Αθήνα. Ε, η απόφαση λαμβάνεται στο Συμβούλιο αλλά με κονδύλια τα οποία θα είναι διαθέσιμα που δεν χρειάζεται κάθε φορά να ε, περνάμε να κάνουμε έρανο για να μαζέψουμε τα χρήματα για μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Κάτι το οποίο βεβαίως θα επισπεύσει πολύ τα πράγματα και υποστήριξη για τους εταίρους. Θα θυμάστε πόσο δύσκολο ήταν να καταλάβουμε ε, πώς θα μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε ε, τις ομάδες ε, στα διάφορα μέρη όπου επενδύουμε για να μπορούν να παραμένουν συμμορφωμένοι με τις συνθήκες αλλά να μπορούν να βοηθούν και σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές για μας όπως το κέρας Αφρικής ή στο Ζαχέλ. Θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Χρησιμοποιούμε ήδη τη διευκόλυνση για την ειρήνη, είναι περιορισμένο θεωρούμε, μόνο στην υποσαχάρια Αφρική. Για ποιο λόγο δεν θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε για παράδειγμα την Τινησία ε, όσον αφορά τη διαχείριση των ε, συνόρων, ε, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, ε, και άλλα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν σε 5-6 χρόνια. Κάποιοι είπαν, ε, συζητούμε τώρα πώς ε, οι διάδοχοί μας θα μπορέσουν το 2026 να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Πρέπει κάπως να σκεφτούμε ένα μέλλον που δεν μπορούμε να το προβλέψουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα κατά πόσο το προσωπικό μας είναι αρκετά πολυσχηδή ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλε αυτέ τι προκλήσει το να υπάρχει ένα μόνο μέσο δεν σημαίνει ότι καταργούμε όλες τις αρμοδιότητες και ότι ε, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν. Προφανώς υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό στην ΕΕΔ, το ίδιο ισχύει και στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έχουμε προσωπικό, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι, έχουν εξαιρετικές δεξιότητες, είναι απολύτως κατάλληλοι και ικανοί και πρέπει να ενθαρρυνθούν να βλέπουν τα πράγματα όχι μόνο μέσα από το πρίσμα ε, μιας γενικής διεύθυνσης συγκεκριμένη ομάδα αλλά λίγο πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Μπορούν να το κάνουν, αλλά πρέπει να του ζητηθεί να το κάνουν, που είναι κάτι που δεν συμβαίνει υποχρεωτικά όταν πρέπει να ασχοληθούν μόνο με ένα συγκεκριμένο μέσο και όχι την ευρύτερη πολιτική. Τώρα, αφιερωμένε ομάδε, ειδικότερα στην πρόληψη των συγκρούσεων, κάποιο το είπε αυτό, μα τι έχουμε ήδη αυτέ τι ομάδε ε, και ίσω θα έπρεπε να ενημερώσουμε ε, τα, τα μέλη του επόμενου κοινοβουλίου σε σχέση με ό,τι ήδη κάνουμε, ίσως θα ήταν χρήσιμο αυτό. Ε, και σοκαρίστηκα που άκουσα ότι ένα συνάδελφο είπε ότι δεν ξέρει πώς δαπανώνται τα χρήματα. Αυτό δεν είναι μόνο δικαίωμά σα, είναι και καθήκον σα να το γνωρίζετε. Οπότε ελπίζω ε, να ε, μπορείτε να ε, εκπληρώσετε αυτό το καθήκον για το οποίο σα ψήφισαν οι ψηφοφόροι σα. Έχετε αυτή την ευθύνη, δεν είναι μόνο δικαίωμα. Είναι ευθύνη να ξέρετε πώ εξοδεύονται τα χρήματα και να κάνετε έτσι τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μήνυμα από πλευρά των διερμηνέων. Σήμερα βρισκόμαστε στην 30η ημέρα ε, διαμάχης με τη διοίκηση και όπως είχαμε ανακοινώσει στην αρχή της συνεδρίασης, η διερμηνία σταματάει στις 4.30 ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Uh, a single instrument helps in this respect because it gives us a strategic coherence to policies, the integrated approach, the global strategy is all about that.